Ε, συνεδρίαση από τις 10 έως τις 1 ε, ε, και το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για το χρόνο που διαθέσατε.